Ντερί, Κάινεμ και Οκτάβια Σάρδο σχετικά με την ε, μεταχείριση των παραγωγών ε, ορνήθων. Έχουν ε, ήδη, έχει ήδη υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία και βάσει του άρθρου 122 του κανονισμού θα μεταδοθεί αρμοδίως με την ένδειξη όλων των ονομάτων που έχουν προσυπογράψει στα πρακτικά. Έχουμε τώρα την, ε, ε, την Σενίσκη Μπεζέ Όνιμπολ Τάκουλα σχετικά με μεγαλύτερη ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, τα, ε, για τον αθλητισμό. Και βάσει του άρθρου 123 και το θέμα αυτό θα δημοσιευθεί στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίας. Ο κύριος Κέλλη μπορεί να μιλήσει για 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε εξ ονόματος όλων των υπογραφώντων <clears throat> του Ιβο Μπαλέτου Χανουτάκουλα, της Μαρίας Χάνεμπολ και άλλων θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Είναι σημαντικό ότι περίπου 50% αυτών που υπέγραψαν ήταν γυναίκες. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ όλους αυτούς που συνεργάστηκαν σε αυτό το εγχείρημα και να αποτίσω ιδιαίτερο <clears throat> φόρο τιμής σε αυτούς οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σημαντικό σε, στην ε, υπογραφή αυτού του ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Γραπτή δήλωση 61 του 2010 υποβληθήσα από τους συναδέλφους Τόμσεν, Λίνε, Φιγερέιδο, Ντέλη και πρώτα Ζιέβιτς. Ο κύριος Ντέλη έχει ζητήσει το λόγο. Πρόκειται για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αστέγους. Ε,